Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη και πάλι για την καθυστέρηση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Μέχρι τις 10 θα εξετάσουμε το σημείο 12 την συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΦΑΟ, αλλά αυτό σε λίγο, γιατί πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που λάβετε όλοι σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν το κοιτάξετε. Η κυρία Χάζεκαμπ μας έστειλε ε, mail ε, την απόφαση των συντονιστών που ελήφθη χθε για την ε, έκθεση για τη μεταφορά των ζώων και την ανάθεση της ε, εκπόνησης σχετικής έκθεσης στην ομάδα μεταρρυθμιστών συντηρητικών. Η κυρία Χάζεκαμπ, από ό,τι κατάλαβα, ε, ήταν ε, η αρμόδια για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, αλλά εξέφρασε σημαντικές επιφυλάξεις και μάλιστα χρησιμοποιεί και μια έντονη διατύπωση στη, στο mail που μας έστειλε. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ανατεθεί αυτή η έκθεση στους ε, συντηρητικούς μεταρρυθμιστές με ψηφοφορία 25 ψήφους υπέρ 17 κατά. Ε, ε, πέντε ε, ψήφισαν υπέρ, από 8, ε, από τους 8 συντονιστές για την ανάθεση στο ECR. Και εδώ δεν ε, χρησιμοποιείται το σύστημα των μόριων. Υιοθετήσαμε μία άλλη μέθοδο. Και αυτό απορρέει από μία προηγούμενη μας απόφαση. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχε και άλλο ενδιαφέρον από άλλη πολιτική ομάδα για την έκθεση αυτή. Και εγώ μάλιστα ε, εντυπωσιάστηκα που αναφέρθηκε ότι έχω τέτοια επιρροή και μάλιστα εδώ αναφέρεται το αίτημα με υπογραφή 20 ευρωβουλευτών ότι εγώ έπεισα τη διάσκεψη των Προέδρων. Και ότι χάρη σε μένα τέθηκε αυτό στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, μα ούτως ή άλλως τέτοια θέματα ή ανήκουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Οπότε δεν χρειαζόταν να γίνει τέτοια ερευνητική προσπάθεια. Όπως ξέρετε, τελικά ανατέθηκε σε εμά αυτή η έκθεση. Με την συμμετοχή ε, και των επιτροπών ΕΜΒΙ και ΤΡΑΝ, περιβάλλοντος και ε, μεταφοράς. Εγώ δεν ήμουν κατά της συμμετοχής ε, των άλλων για γνωμοδότηση, παρόλο που κάτι τέτοιο αναφέρεται στην επιστολή. Δεν θέλω να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Στεναχωρήθηκα. Ούτως ή άλλως η κυρία Χάζεκα μπορεί να είναι σκιώδη ηγετήρια στην έκθεση και να συμβάλλει στη διαμόρφωση της έκθεσης. Ξέρουμε πόσο ικανή είναι η κυρία Χάζενκαφ, πόσο ασχολείται με τα θέματα αυτά, με τη θέρμη τα εξετάζει και τι τεράστιες γνώσεις έχει για το θέμα αυτό της μεταφοράς των ζώων και πόσο αφοσιωμένη είναι στο ζήτημα της προστασίας των ζώων και της ευζοίας οπότε θα μπορέσει ούτως ή άλλως και ως και να συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου της έκθεσης και να την τροποποιήσει και με την υποβολή τροπολογιών. Ε, λυπάμαι αν ε, δόθηκε εντύπωση ότι εγώ παρενέβη στο έργο της Επιτροπής. Ε, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά πραγματικά δεν έγινε σε καμία περίπτωση εσκεμένα. Και νομίζω ότι πραγματικά ήταν λίγο υπερβολική η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην επιστολή, αλλά καταλαβαίνω, ήταν μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, γι' αυτό ήταν λίγο υπερβολική η διατύπωση. εγώ νομίζω ότι το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξεν. Υπάρχει λιμένη απόφαση των συντονιστών. Αυτά λείπουμε για αυτή την εισαγωγή που χρειάστηκε να κάνω, αλλά έκρινα σκόπιμο να, κάνω, να δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Τώρα, περνάμε σε άλλο θέμα. Έρχονται κάποιες στιγμές που προκαλούν μια θλίψη, όπως τώρα, και δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτά τα θέματα, γιατί αποχωρεί ένα συνάδελφο με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Μιλάω για τον κύριο Ζαμπόλ Ντενανό, που αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί στα τέλη του μήνα. Αποφάσισε να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί έκρινε να αποχωρήσει. Μια χαρά μου φέρεσε, ακμεότατος. είσαι σε μεγάλη φόρμα, έχεις συντάξει πολύ άρτιες και αξιόλογες εκθέσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος δεν έλαβε μία απόφαση, οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Ήταν και προηγουμένω ε, για μια σύντομη περίοδο Ευρωβουλευτή και μετά τι τελευταίε εκλογέ από το 2014, αλλά έχει μακρά σταδιοδρομία στην ε, περιφέρεια Λιμουζά στη Γαλλία. Και το μεγαλύτερο ρυθμό της ζωής του το πέρασε ε, σε διάφορα μέρη εργαζόμενος. Ξεκίνησε το 1987 τη σταδιοδρομία του, ε, διετέλεσε αντιδήμαρχος, δήμαρχος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Λιμουζά. Φαίνεται ότι ε, αγαπάει πολύ την πατρίδα του, γι' αυτό και μεγάλο τμήμα της ζωής το πέρασε εκεί απασχολούμενος ε, σε διάφορα ε, σημεία και σε διάφορες θέσεις. Επίσης, ήταν ε, πολύ ενεργό μέλος της Επιτροπής Άγκρη και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θυμάμαι την τελευταία του έκθεση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες. Και ήταν πολύ συμπαθής συνάδελφος η παρουσία του μας χαροποίησε. Αλλά έχω ένα παράπονο, κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Ντενανό. Έχω ένα μεγάλο παράπονο απέναντι σας. Γιατί ξέρω ότι είστε πολύ παθιασμένος και έχετε σημαντικές επιδόσεις ως μουσικός. Παίζετε κιθάρα και ακορντεόν. Και μάλιστα είστε γνωστός, διάσημος στη Γαλλία για το μουσικό σας ταλέντο Μάλιστα διακριθήκατε στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην Προέδρου Φρανσουά Ολάντ το 2012. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια δική σας παράσταση, ενα μείνει κονσέρτο. Μακάρι να μας κάνετε αυτή την τιμή, είτε εν ώψη των εορτών, είτε σε κάποια άλλη ευκαιρία να μας δώσετε μια μήνυ συναυλία, να μας παίξετε λίγο ακορντεόν για να έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε. Γιατί είναι ωραίο να έχει κανείς πάθη και ιδιαίτερα να έχει ως πάθος τη μουσική. Ένα μουσικό ταλέντο το εκτιμώ ιδιαίτερος γιατί εγώ δεν έχω κανένα απολύτως ταλέντο στη μουσική. Δεν έχω μουσικό αυτή. Και αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Ακόμη και στις γλώσσες. Ε, δεν έχω μουσικό αυτή, είμαι παράφωνος, δεν μπορώ να τραγουδήσω, γι' αυτό και με εντυπωσιάζουν πολύ όσοι ασχολούνται με τη μουσική. Η σχέση μου με τις νότες και μου τη μουσική είναι πολύ α, δυσάρεστη δυστυχώς. Σας ζηλεύω πραγματικά. Με θετικό τρόπο φυσικά. Αλλά πραγματικά σας θαυμάζω πολύ. Κρίμα που δεν είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια συναυλία σας με ακορδόν Σας εύχομαι πάντως ε, καλή τύχη στη συνέχεια και αν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο, πολύ ευχαρίστως. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Εσείς κύριε Ντενανό, αποχωρείτε τώρα, άλλοι θα αποχωρήσουμε μετά τις εκλογές δεν θα επανεκλεγούμε και θα γυρίσουμε στις πατρίδες μας πολύ από εμά όπως και εσείς τώρα. Αυτά και αν θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ. Αυτή είναι η στιγμή. Ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ πρόεδρε για τα λόγια σας που ήταν δίκαια και εύστοχα και πολύ θερμά και ανθρώπινα. Πραγματικά ανταποκρίνονται στην προσωπικότητα του Ζαν Και θέλω εδώ συντονιστής και φίλος από πλευράς μου, φίλος και συντονιστής σε αυτή τη σειρά, είναι πιο σωστή, να πω πόσο χάρηκα που είχατε δυνατότητα να συνεργάζομαι με τον Ζαν Πολντενανό. όπω είπατε, πέραν τον, ε, του χαρίσματός του ως μουσικού, που το επιβεβαιώνω, είναι από αυτούς τους μεγάλους πολιτικούς άνδρες που ανακάλυψα κάπως καθυστερημένα, το αναγνωρίζω, όμως για τον οποίο ο ορισμός της αφοσίωσης, της πίστης, του ανθρωπισμού και εργατικότητά του είναι λέξεις κλειδιά της καθημερινής του ζωής. Και θέλω εδώ να προσθέσω και την έννοια του σεβασμού. Διότι είναι μέρος αυτής της πανοπλίας με την οποία ε, ήρθε να εργαστεί εδώ ο κύριος Δενανό σε έναν τομέα ε, κυρίω των αγροτικών, ε, τον οποίο εργάζεται, και στον κόσμο της υπαίθρου. Αφορά ιδιαίτερα πολλούς πολιτικούς άντρε και η Γαλλία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Στο Λιμουζά ε, μας απασχολούν τα θέματα αυτά Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι βρίσκεται στην καρδιά των προβληματισμών του κυρίου Ντενανό και στο κέντρο της πορείας του. Πραγματικά το θέμα της επαφής με το κοινό, ε, της αφοσίωσης, της δημοκρατικότητας, ε, της πίστης του, ε, είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλη του την επαγγελματική σταδιοδρομία και ήθελα και εγώ από πλευράς μου να τον ευχαριστήσω που είναι αυτός που είναι, καταρχάς και έπειτα για όσα ε, πέτυχε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομία. Το λέω πέραν κάθε επισημότητας με απόλυτη βαθιά φιλία. Είναι ένας πραγματικός πολιτικός άντρα, τον ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να δώσω ε, αυτό το χαιρετισμό με τροποφιλικό ε, στον κύριο Ντενανό. Να πω αυτά τα λίγα λόγια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντριώ, κύριος Ντάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Σινκέρσκι και τον Έρικ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας μας για την εξαιρετική συνεργασία. Να ευχηθώ καλή κάθε επιτυχία στην συνέχεια σε ό,τι κάνετε Ελπίζω κάποια στιγμή να μας ξανάρθεις και, και εξ ονόματος της ομάδας μου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς είμαι βαθιά συγκινημένος με αυτά που γίνονται σήμερα το πρωί, με το άνοιγμα αυτής που είναι για μένα η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για αυτές τις στιγμές που για μένα είναι ιδιαίτερες. Το παραδέχομαι. Πρόεδρε, πραγματικά εκτίμησα ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύσατε σε αυτή την Επιτροπή και για το κύρος σας και για την καλοσύνη με την οποία εξυπηρετήσατε τη λειτουργία αυτή τη επιτροπή Είναι πολύ σημαντικό. Και ευχαριστώ και του συναδέλφου για το σεβασμό του. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Σεβασμό μεταξύ των μεν και των δε. Ο καθένα μπορεί να εκφράσει τι απόψει του όπως νομίζει στην Επιτροπή αυτή. Ο καθένα δίνει τι ιδέε του, εκθέτει τι ιδέε του και μετά μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια σύνοψη και να συνδυάσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη γεωργία της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά της Ευρώπης και της Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων. Ότι προσπαθούμε να ε, ανακεφαλαιώσουμε και να συνδυάσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Από μένα λοιπόν ε, μια έκφραση σεβασμού και πολλές ευχαριστίες για όσα κάνατε και μπορεί να μην έρθω σίγουρα με το ακορντεόν όμως θα ξανασχοληθώ με την ε, μουσική σοβαρά, διότι εδώ και τέσσερα χρόνια με τη θητεία μου ε, εγκατέλειψα λίγο την ε, πορεία μου. Πάντως, πέρα από τη μουσική, δυστυχώς δεν κατάφερα να μάθω αγγλικά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μου απογοήτευση αυτά τα χρόνια προφορά των αγγλικών δεν μου πάει, αλλά στη μουσική θα συνεχίσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ όλους σας. Σας ευχαριστούμε. Merci μποκού. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ξέρετε, έλαβε χώρα το Παγκόσμιο ε, Συμπόσιο για το έδαφος 2 με 4 Μαΐου στη Ρώμη, στα κεντρικά γραφεία της ΦΑΟ. Ε, δεν μπορέσαμε να λάβουμε μέρος γιατί είχαμε και τη μήνυ ολομέλεια. Ε, δεν ξέρω αν κάποιος μπόρεσε να πάει. Πάντως ζητήσαμε από εκπροσώπους της ΦΑΟ να έρθουν για να μας ενημερώσουν για την έκβαση αυτού του συμποσίου και επειδή για λόγους υγείας ο κύριος Βάργας δεν μπόρεσε να παραστεί, αντικαθίσταται από τον κύριο Ροντρίγκο Ντελα Πουέρτα και την κυρία Νατάλια Ευγένιο από τη Γενική Γραμματεία ε, για την καταπολέμηση της ρήπανσης του εδάφους. και από το Γραφείο Σύνδεσης ε, το, της ΦΑΟ της Βρυξέλλες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί η ποιότητα του εδάφους ε, επηρεάζει ολόκληρο το περιβάλλον. Και φυσικά την παραγωγή τροφίμων. Το θέμα της διαχείρισης ε, των εδαφών είναι πολύ σημαντικό γιατί μειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο οι γεωργικές εκτάσεις, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε ποιοτικά εδάφη. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να μας κάνουν την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Τελαπουέρτα, κυρία Ροντρίγκες Εουζένιο. Θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση μετά την παρουσίαση των δύο εμπειρογνωμόνων. Πάντως χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία εδώ των εκπροσώπων της ΦΑΟ, γιατί τιμούμε ιδιαίτερο στη στενή συνεργασία που έχουμε με τη ΦΑΟ, γιατί έχουμε κοινού στόχους με την οργάνωση αυτή. Παρακαλώ. Ε, thank you very much, Honorable Chair. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλημέρα σας. Με χαρά μου σήμερα θα σας μιλήσω για τα υγιή εδάφη και την συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και την Γεωργία. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που αποδίδεται στο ζήτημα των εδαφών. Θα θυμάστε τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή αυτή μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης είχε μια σειρά συζητήσεων και συνεδριάσεων επευκαιρία του Διεθνούς Έτους Εδαφών και της Διεθνούς ημέρας Εδαφών. Κυρίε και κύριοι, τα εδάφη είναι το θεμέλιο της Γεωργίας και το μέσο στο οποίο αναπτύσσονται όλα τα καρποφόρα φύτα. 95% των τροφίμων που τρώμε άμεσα ή έμεσα παράγεται από τα εδάφη. Τα υγιή εδάφη είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για την ε, τροφική αλυσίδα. Παρέχουν ε, τα θρεπτικά στοιχεία το νερό και το οξυγόνο που χρειάζονται τα φυτά. Βεβαίως όταν ε, μολυνθούν μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα περισσότερα εδάφη είναι σε κατάσταση καλή ή, κακή, ή πολύ κακή και η κατάσταση θα μπορούσε να χειροτερέψει αν δεν αναλάβουμε δράση σε όλα τα επίπεδα, το κρατικό, το ατομικό, το κοινοβουλευτικό, σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. Η ρήπανση των εδαφών ε, είναι κάτι το οποίο έχουμε παραμελήσει ε, επί σειρά ετών, ε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται με γυμνό μάτι. Είναι κάτι το κρυφό. Ε, αντιλαμβανόμαστε τη ρήπανση στον αέρα, στο νερό, δεν αντιλαμβανόμαστε την ρήπανση των εδαφών. Τα εδάφη δρούν ως ε, φίλτρο των ρήπων για να μην μπουν στο διατροφικό σύστημα. Υπάρχει όμως και ένα όριο στις δυνατότητες τους ε, να αντιμετωπίσουν την ρήπανση. Η σοδαφών μειώνει την ποιότητα του νερού, του αέρα και έχει και οικονομικό κόστος. Ε, υπονομεύει την ασφάλεια τροφίμων, καθώς πέφτει η στρεματική απόδοση και γίνονται πλέον ακατάλληλα τα τρόφιμα για κατανάλωση. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι οι βασικές αιτίες της ρήπανσης. Οι βιομηχανικές και αστικές δραστηριότητες απελευθερώνουν μεγάλους χημικών ουσιών, σκουπιδιών στο περιβάλλον και το ίδιο ισχύει και για την ίδια γεωργία και εκτινοτροφία. Οπότε η πρόληψη της ρήπανση ε, των εδαφών θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα παγκοσμίω. Ο Οργανισμός ε, Τροφίμων και Γεωργίας ε, είναι προσιλωμένος στην βιώσιμη διαχείριση των εδαφών και στα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η ρήπανση των εδαφών. Το Παγκόσμιο Συμπόσιο για την ε, ρήπανση των εδαφών που ανέφερε ο πρόεδρος έλαβε χώρα πριν 15 μέρες ε, στην ε, Ρώμη με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε συνεργασία πολλών εταίρων και συγκεντρώθηκαν επιστήμονες, η τεχνολογική κοινότητα, οι γεωκτήμονες ε, και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση. Και βεβαίως ακριβώς έχουμε το θέμα που υπάρχει και στην ε, δική μας ε, τη χώρα και σε γειτονικέ χώρες που μας παρέχουν με διάφορα αγαθά. Είναι, γνω... είναι άγνωστο Λοιπόν, ποιο είναι ο βαθμό τη ρήπανση των εδαφών, γιατί κυρίως μιλάμε για αναψώμενες χώρες που δεν έχουν τους πόρους και τι δυνατότητε να αξιολογήσουν και να διορθώσουν την κατάσταση. Ο οργανισμός μας ε, πράγματι βοηθάει τις χώρες που χρειάζονται αυτήν την βοήθεια και αυτή τη στιγμή διεξάγει μια συνολική αξιολόγηση της ε, ρήπανσης ε, των εδαφών. Η επιστημονική βάση, όπως θα εξηγήσει και η συνάδελφος, η κυρία Ροντρίκες, είναι σαφής. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Θα ήθελα τώρα, επί τη ευκαιρία, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την στήριξή της στην παγκόσμια αυτή συνεργασία για τα εδάφη για το έργο του οργανισμού μας για τα υγιή εδάφη. Ελπίζουμε η συνεργασία μας αυτή να αυξηθεί στο προσεχές μέλλον. Και βεβαίως ε, γεγονός είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποιον ρόλο να παίξει. Συναδελφός μου, η κυρία Ροντρίγκε Σονχένιο, επίσης από την Ισπανική Μαφία, από την ε, Παγκόσμια Γραμματεία του Εδάφους, θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση για τα ευρήματα και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Rodrigo, for... Ευχαριστώ πολύ, Ροντρίγκο, για αυτή την εισαγωγή. Μας ε, ενέπνευσε η ομιλία σου. Θα σας παρουσιάσω τις τεχνικές πτυχές της ε, ρήπανσης των εδαφών, προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσω τα βασικά μας πορίσματα, της συστάσεις από το συμπόσιο. Ο Ροντρίγκο ανέφερε ότι η ρήπανση των εδαφών είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι εμφανής. Γιατί, γιατί υπάρχει χημική φθορά. Υπάρχουν ουσίες σε μεγάλη συγκέντρωση που πέραν του φυσιολογικού συγκεντρώνονται στα εδάφη. Το διακυβερνητικό παγκόσμιο πάνελ για τα εδάφη, ε, το τεχνικό μας πάνελ, μέσω της εταιρικής μας σχέσης, εκπώνησε αυτή την έκθεση το 2015 για τις βασικές απειλές στα εδάφη, κατά των εδαφών και το, της υγείας. Η ρήπανση των εδαφών λοιπόν ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες ε, ρήπανσης. Στην Ευρώπη και την Ευρασία η ε, ρήπανση των εδαφών είναι ο τρί, τρίτη πηγή κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Εμείς είμαστε οι βασικοί υπεύθυνοι για αυτή τη ρήπανση, οι ανθρώπινες δραστηριότητε. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, μεγάλος αριθμός ε, επικίνδυνων συστατικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. 144.000 χημικές ε, ουσίες κάθε μέρα ε, εκλείονται, απορρίπτονται στο περιβάλλον. Ε, και δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους σύσταση. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουμε πάνω από 340.000 ε, σημεία που έχουν ε, ήδη πληγεί από τη ρήπανση αυτή και θα χρειαστούν αποκατάσταση. Κάτι που επιφέρει μεγάλο κόστος βεβαίως. Οι εκτιμήσεις λένε ότι 2,8 εκατομμύρια σημείων μπορεί να έχουν παρόλα αυτά πληγεί από την συγκεκριμένη ρήπανση στην Ευρώπη και μόνο. Επιπλέον δεν γνωρίζουμε το βαθμό της ε, διάχυτης ρήπανσης των εδαφών που κυρίως ε, οφείλεται στην χρήση των ε, χημικών ουσιών για, για γεωργικούς σκοπούς. Η ρήπανση των εδαφών, όπως είπε και ο Ροντρίγκο και ο πρόεδρός σας, έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού, την ατμοσφαιρική ποιότητα, αλλά και τον δείκτη για την υγεία μας, το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την παραγωγή τους ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι 9 δις ε, άνθρωποι μέχρι το 2050 υπολογίζεται. Και βεβαίως ε, θα βασίζονται στην ε, ασφάλεια των τροφίμων, τα υγιεινά τρόφιμα. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών, ώστε να βελτιώσουμε την παραγωγή τροφίμων κατά 58% ε, για τον προβλεπόμενο ανθρώπινο πληθυσμό που θα χρειαστεί όμως 60% αύξηση στην παραγωγή των τροφίμων ε, σε αντίθεση με το 58% που σχεδιάζουμε. Εάν εφαρμόσουμε λοιπόν τις πρακτικές βιώσιμες διαχείρισης των εδαφών μπορεί και να τα καταφέρουμε. Η ρήπανση των εδαφών είναι μια πραγματική απειλή και κατά των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχων που όλοι δεχτήκαμε και εγκρίναμε. Η επίτευξη των 12 στόχων συνδέεται απευθείας με την πρόληψη και την, ε, τον περιορισμό της ρήπανσης των εδαφών. Το Παγκόσμιο Συμπόσιο για τη ρήπανση των εδαφών ε, είδαμε ότι υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Συγκεντρώσαμε πάρα από 500 επιστήμονες, πολιτικούς υφήνοντες, ανθρώπους από τις επιχειρήσεις, από τις κυβερνήσεις και αυτών που εργάζονται στην πράξη με τα εδάφη. Είχαμε ένα τριήμερο εντατικών εργασιών, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις που θα σας παρουσιάσω τώρα. Είναι σαφές ότι η ρήπανση των εδαφών είναι μια απειλή παγκοσμίω. Είχαμε παρουσιάσεις από όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του συμποσίου και βλέπετε σε αυτό το γράφημα παντού ότι αντιμετωπίζεται το ίδιο πρόβλημα. Μας ανησυχεί αυτό, αλλά έχουμε επιτέλους μια ευκαιρία. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, η τελευταία συνέλευση της, ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον υπέγραψε μια σχετική, ε, μια σχετική δήλωση για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της ρήπανσης των εδαφών. Τα βασικά συμπεράσματα του συμποσίου λοιπόν ήταν ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικός ότι η ρήπανση των εδαφών είναι πραγματικά μια ε, σοβαρή απειλή για την παραγωγικότητα της γεωργίας, την ασφάλεια των τροφίμων και την ανθρώπινη υγεία ότι η αντιμετώπιση της ρήπανσης των εδαφών απαιτεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και δική σας συμμετοχή όλων μας εδώ για να προλάβουμε να ε, ελαχιστοποιήσουμε και να αποκαταστήσουμε τα εδάφη. Οι βασικές πηγές ρήπων προέρχονται από τις ανθρωπογενείς δράσεις. Η βιομηχανία, ο βιομηχανικός κλάδος, οι εταιρείε, η αποκομιδή λιμάτων ή γεωργία. Πρέπει να περάσουμε σε βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των εδαφών. Η πρόληψη της ρήπανσης των εδαφών θα πρέπει να γίνει μια κορυφαία προτεραιότητα παγκοσμίω, διότι το κόστος για την αποκατάσταση των εδαφών που έχουν ρηπανθεί είναι τεράστιο. Γι' αυτό λοιπόν η πρόληψη θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα κάνουμε η κατάσταση του φαινομένου της ρήπανσης των εδαφών παγκοσμίω ακόμα δεν έχει καταγραφεί πλήρως. Βασιζόμαστε σε εθνικά συστήματα πληροφοριών και πρέπει βεβαίως ως προϋπόθεση να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας για να αντιμετωπίσουμε, να βρούμε λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε πιλωτικές μελέτες σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ιδίως στην Αφρική και την Ασία, διότι εκεί θα έχουμε τα περισσότερα προβλήματα είναι πολύ αδύναμες οι νομικές δυνατότητες για τον έλεγχο της ρήπανσης των εδαφών και δεν έχουμε καθόλου δεδομένα για το τι συμβαίνει εκεί. Οι συστάσεις των ε, συμμετεχόντων που συμφωνήθηκαν από όλους στο συμπόσιο είναι ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε ε, από τα παιδιά και τους νέους ως τους πολιτικούς ηθήνοντες, αυτούς που είναι χρήστες των εδαφών στην πραγματικότητα, που ασχολούνται στην πράξη με τα εδάφη, να δουν ε, περί τίνος πρόκειται και πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, πώς μπορεί να υπάρξει πρόληψη και αποκατάσταση. Ο ε, ρόλο τη παγκόσμια εταιρική σχέση για τα εδάφη και τη ρήπανση των εδαφών είναι σημαντικός. Έχουμε εκστρατείε ευαισθητοποίησης κάθε χρόνο για τις βασικέ απειλέ κατά των εδαφών. Φέτος ε, και πάλι θα οργανώσουμε μία ε, εκστρατεία ευαισθητοποίηση, ιδίω την, ημέρα για την Παγκόσμια Μέρα για τα Εδάφη το Δεκέμβριο. Θα σα πω περισσότερα αργότερα. Και άλλη μία ιδέα που προέκυψε από το συμπόσιο ήταν να οργανώσουμε δύο τεχνικές ομάδες εργασίας για να προσφέρουμε στοιχεία για μια τεκμηριωμένη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θα χρησιμοποιηθούν κατευθυντήριες γραμμές που θα ενταχθούν στο σωστό πλαίσιο για την αποτίμηση τον έλεγχο και την καταγραφή των φαινομένων ρήπανση των ανταφών. Όπω είπα, η πρόληψη τη ρήπανση των ανταφών. άμεση Θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα για να προλάβουμε πρέπει να εφαρμόσουμε τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές όπως τον κόντεξ ελιμετάριους, της ΦΑΟ, τις ε, ε, εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση των εδαφών, όσα ισχύουν τον κώδικα συμπεριφοράς για τα φυτοφάρμακα και τη διαχείρισή τους, το ε, παγκόσμιο πλάνο και Ίσως έτσι σε έναν βαθμό να πετύχουμε κάποια πρόληψη και επίση πρέπει να ενισχύσουμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων και τι δραστηριότητε εκπαίδευση για την πρόληψη της ε, ρήπανση των εδαφών. Όπως σας είπα προηγουμένως θα ξεκινήσουμε μια σημαντική εκστρατεία ευαισθητοποίηση στην Παγκόσμια Μέρα για τα εδάφη το Δεκέμβριο και αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε και να, συμμετάσχετε και να ε, χρησιμοποιήσετε το hashtag Soil Pollution, ε, ρήπανση των εδαφών. Φέτος θα εκδώσουμε μάλιστα και το, τα έγγραφα ε, που προέκυψαν από το συμπόσιο προσπαθώντας να επιδιώξουμε και θα επιδιώξουμε την εφαρμογή των συστάσεων υπάρχουν και τεχνικά εγχειρίδια τα οποία εκπονούμε τώρα για την ε, ρήπανση των εδαφών την αποκατάσταση και την εξέβρεση λύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, σε συγκεκριμένε περιοχέ του κόσμου. Όμω έχουμε και σοβαρού περιορισμού. Χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερου πόρου για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε συγκεκριμένε δράσει και να βοηθήσουμε να βρεθούν λύσει για τα εδάφη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να αποτιμήσουμε φοροτιμή τη δουλειά και την προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μα στηρίξει, όμω πρέπει να συνεχίσετε. Η ρήπανση των εδαφών είναι μια απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μπορεί μόνο να ε, αντιστραφεί εφόσον υπάρξει δράση ε, ε, στην πράξη. Πρέπει λοιπόν όλοι να εργαστούμε για την αποκατάσταση των εδαφών και την ασφάλεια των τροφίμων. Τώρα έχουμε ήδη κάποιε πρώτε κινήσει, επιστημονικά στοιχεία και δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίε. Είναι καιρό για δράση. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε. Ζήτησαν το λόγο η κυρία Σάρα, ο κύριος Βάιτς, ο κύριος Χόισλινγκ. Παρακαλώ πολύ σύντομα ένα λεπτό, γιατί στις 10 θα αρχίσουμε τη δημόσια ακρόαση από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κυρία Σένερα, παρακαλώ ένα λεπτάκι, όχι παραπάνω. Θερμή παράκληση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας για την παρουσίαση της έκθεσης της ΦΑΟ. Πολύ σημαντική έκθεση. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα, τη Γαλλικία, όπου σημαντική, ε, μια από τις σημαντικές δραστηριότητες που έχω και ευρωβουλευτής είναι να επισκέφτομαι ε, περιοχές στην Ήπεθρο που έχουν επηρεαστεί από την κακή διαχείριση αποβλήτων, βιομηχανικών λιμάτων και ε, αποβλήτων πάσης φύσεως. Γιατί οι αυτόνομες ε, ε, περιφέρειες της ε, Ισπανίας χρησιμοποιούν εγκαταλελειμμένους χώρους και εγκαταλελειμμένους χωματερές για να θάψουν απόβλητα από όλη τη χώρα και μάλιστα με πολύ κακή διαχείριση των αποβλήτων. Ε, αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο γιατί αυτοδηλητηριαζόμαστε, δηλητηριάζουμε τα εδάφη μας και δηλητηριάζουμε τον αγροτικό μας πληθυσμό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και είναι σημαντικό να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα. Γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος, θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει και στην Επιτροπή Γεωργίας. Για να δούμε αν αυτό το φαινόμενο συμβαίνει μόνο στη, ε, στη δική μου χώρα, την Ισπανία, ή είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο αυτή η άκρητη διαχείριση αποβλήτων οπουδήποτε και χωρί μέτρα προστασία. Ευχαριστώ. όντω. θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο θέμα αυτό στην Επιτροπή. Ο κύριος Βάιτς, θα είμαι πολύ σύντομο. Θα πρέπει να αλλάξει η παρούσα κοινή γεωρική πολιτική ώστε να λαμβάνει υπόψη περισσότερο την προστασία των εδαφών. Ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Άλλε χώρε εφαρμόζουν πιο εκτεταμένη αγρανάπαυση και μάλιστα μερικέ φορέ αγραναπαύουμε πολύ χρήσιμο γεωργικό έδαφο περίεργες επιφάνειες. Βέβαια, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και τον ψεκασμό ή να χρησιμοποιήσουμε drones. Πρόκειται για νέες τεχνολογίες, ακριβίας. Τι γνώμη έχετε για αυτά. Μόσες, Ο κύριος Χόιτεμα. Ευχαριστώ. Ε, όπως και ο κύριο Άγγινιο χρειάστηκε να πάω σε άλλη επιτροπή για να ψηφίσω και δεν παρακολούθησα από την αρχή την ε, παρουσίαση της μελέτης ε, του συμποσίου, των πορισμάτων του συμποσίου. Πάντως είναι πολύ χρήσιμο αυτό το θέμα και σίγουρα η καλύτερη ποιότητα του δάφους έχει τεράστιο δυναμικό και βελτιώνει και την κατάσταση στη γεωργία, εξασφαλίζει πιο βιώσιμη παραγωγή επηρεάζει και την ποιότητα του ύδατος, αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και σίγουρα πιο καινοτόμε τεχνολογίε σε συνδυασμό με οικολογική τεχνολογία θα συμβάλλουν στη βελτίωση τη ποιότητα του εδάφου. Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για τον κανονισμό για τα λοιπάσματα. Και εκεί έχουμε μια πρόταση για τη μείωση των, των ποσοστών καδμίου στα τεχνητά φωσφορούχα λοιπάσματα. Εγώ είμαι υπέρ αυστηρών οριακών τιμών καδμίου, γιατί κάτι τέτοιο συνάδει με την ποιότητα του εδάφους. Βέβαια, δεν θα κατηγορήσουμε αν υπάρχει πολύ κάδμιο στο έδαφος ε, την ε, βιομηχανία παραγωγής τεχνητών λοιπασμάτων, αλλά το γεωργό. Ε, δεν θεωρείτε ότι αυτή είναι καλύτερη στιγμή για να έχουμε πιο αυστηρή νομοθεσία για τα τεχνητά λοιπάσματα και την περιεκτικότητά του σε κάδμιο. Τι γνώμη έχει φάω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ σύντομα να απαντήσετε γιατί ε, καταφθάνουν τα μέλη της Επιτροπής περιβάλλοντος για την κοινή αυτή δημόσια κρόση. Βέβαια καλό θα ήταν να ακούσουν αυτά που θα πείτε γιατί είναι σημαντικό και για το περιβάλλον ε, το ζήτημα της ποιότητας των εδαφών. Κύριε Φλάναγκα, αν θέλετε το λόγο παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. Μια από τις βασικές μου μέρες όταν ήθελα να εκλεγώ εδώ ως Ευρωβουλευτής δεν ήταν ότι θα έρχομαι εδώ για να τοποθετούμε πάρα πολύ γρήγορα επειδή δεν προλαβαίνουμε στο χρόνο που μας αναλογεί. Τέλος πάντων, ε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλο που δεν ήταν εδώ πάρα πολλοί κόσμος στην αρχή της, ε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Θα ήμασταν κρύα τα εδάφη, δεν ήταν υγιή. Είναι κρίμα που ήμασταν τόσο λιγάριθμοι στην αίθουσα λοιπόν. Λες και σίγουρα συμβαίνουν και άλλα πράγματα στον κόσμο, αλλά ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Άγνιου Βεβαίως υπάρχουν ωφέλη από την αναεροβική ε, χόρνευση και την ε, λιματολάσπη, την, ε, τον καθαρισμό της, όμως πρέπει να σκεφτούμε τις σοβαρές ανησυχίες για το τι γίνεται με την λιματολάσπη πριν την αποκαθαρίσουν, δηλαδή το κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα, και βλέπω εδώ ένα κεφάλαιο στο εγγραφό σας για το θέμα αυτό. Πόσο πολύ έχει απασχολήσει και πόσο μπορούμε να ε, κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την κατάσταση ε, και που έχουν γίνει σφάλματα. Τι μπορεί να γίνει με την ε, δασοκομεία επίσης. Και παρόλο που είμαι ευφυές ίσως ζω, φοβάμαι ότι πηγαίνουμε στο δρόμο του ε, σκουλικιού ε, που ε, όπως κάναμε και στο πείραμα του σχολείου βάζαμε ένα σκουλίκι στο βάζο με το χώμα που ανακάτευε όλες τις τρώσεις. Νομίζω ότι το ίδιο κάνουμε όσοι λύθοι. Αν δεν ε, ε, ε, ασχοληθούμε να το συζητήσουμε μεταξύ ξενοτών. Τέλος πάντων αυτό που γίνεται εδώ είναι μια φάρση.